Έχω λάβει την τοποθέτηση του Συμβουλίου για την πρώτη ανάγνωση, την διαιτιολόγηση σχετικά με ε, την ε, δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ε, την σήμανση της Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς και ε, αύριο αρχίζει η προθεσμία μέχρι τις 16 ε, Σεπτεμβρίου για την υποβολή τροπολογιών. Σχετικά ε, με την Λευκορωσία δίνω το λόγο στην κυρία Ντεκάιζερ για να κάνει μια σημαντική δήλωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε για αυτή την διακοπή αλλά θα ήθελα να κάνω μία έκκληση πριν αρχίσω να ασχολούμαι με την περίπτωση της Ράφα Ναζέτ που είναι μία ε, ε, Σύρια ψυχαναλίστρια η οποία συνελήφθη στο Παρίσι την ώρα που πήγαινε να παρασταθεί στον τοκετό της κόρης της και έκτοτε δεν έχουμε νέα της και αν δεν ανακοινωθεί επισήμως το όνομά της οι άνθρωποι εξαφανίζονται και σκοτώνονται. Οπότε σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να κάνω αυτή την έκκληση καταρχήν. Ωραία. Τώρα μπορούμε να αρχίσουμε με τη Λευκορωσία ε, την περίπτωση του κυρίου Μπιαλάσκη ε, και δίνω τον λόγο στον κύριο Ρωμέ Βερουέντα. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να μιλήσουμε όντως για την ε, Λευκορωσία που μας απασχολεί πολύ το θέμα συλλήψεων που γίνεται σε βάρος υπεραπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συμφωνήσαμε στο ψήφισμα αυτό ότι θα υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι οι αρχές της ε, Λευκορωσίας επωφελήθηκαν από τη διεθνή συνεργασία και οικονομικά ε, με βοήθεια της Πολωνίας, τη Λιθωνίας κλπ. Με τις διάφορες όμως πιέσεις, εμείς αυτό που θέλαμε ήταν να βρεθούν τρομοκράτες, αλλά η χώρα το χρησιμοποίησε για να ελέγξει τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και να ενισχύσει τη θέση της. Κάτι που είναι σε βάρος της κοινωνίας των πολιτών και κάτι που καταδικάζουμε. Και λυπούμαστε πάρα πολύ που έτσι ανεύθυνα ε, συμπεριφέρθηκαν οι δημοσιονομικές αρχές της Πολωνίας και της Λιθουανίας. Το ψήφισμα αυτό καταδικάζουμε επίσης την συνεργασία που γίνεται με την Τράπεζα της Σκωτίας και με κάποιες άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Το καθεστώς του Λικοσέκο δεν μπορεί να αποφελείται από τέτοιες συμφωνίες. Είναι πολύ σοβαρό. Και είναι αλήθεια ότι έχουν πάρει την απόφαση τελικά να απάψουν τέτοιες δραστηριότητες. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε έκκληση σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες και δημοσιονομικούς οργανισμούς να σταματήσουν κάθε οικονομική συνεργασία με τις αρχές της Λευκορωσίας. Και υποφελούμε από την ευκαιρία αυτή για να σας το θυμίσω αυτό και να μην συνεχίσουμε τη δουλειά μας αν να μην συμβαίνει τίποτα όπως κάνουμε συχνά με τέτοιες περιπτώσεις δικτατορικών καθεστώτων. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τάνοκ, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή κατάσταση στη Λευκορωσία είναι αξιοθρύνητη. 20 χρόνια μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, το γεγονός ότι ο Λουκασέγκο μέχρι στιγμής, μέχρι τη σήμερον ημέρα και ε, παρά τις ε, ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις χρησιμοποιεί την βία για να καταστήλει υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαράδεκτο. Επίσης τα αποτελέσματα των δίθεν εκλογών πέρσι ήταν ε, εξίσου αξιοθρύνητα θα πρέπει λοιπόν εμείς ε, σε όλες τις ε, πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες να επιμείνουμε ότι θα πρέπει να επικρατήσει η δημοκρατία και να μπορέσουν να μπουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια που ανήκουν. γενικά το κοινό της Λευκορωσίας είναι έτοιμο για να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά για να γίνει μια τέτοια μετάβαση το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι ισχυρό και ενωμένο. Η ECR πιστεύει ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μα με τη δημοκρατική αντιπολίτευση για να ενισχύσουμε μια αίσθηση κοινή λογοδοσία αλλά πρέπει να δείξουμε και τις δράσεις μας, να ενισχύσουμε τις δράσεις μας με επικυρώσεις κατά του καθεστώτος, ώστε να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ζητάμε λοιπόν από ολόκληρη την κοινότητα να παγώσει την οικονομική βοήθεια προς το καθεστώς μέχρι ισότου όλοι όσοι έχουν ε, συλληφθεί παράνομα, οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως ο Μπιαλάτσχη, ε, δημοσιογράφοι καθώς και προεδρικοί υποψήφοι να απελευθερωθούν και να αρθούν οι κατηγορίες εναντίον τους. Ε, η Λευκορωσία είναι μια χώρα με πολιτισμένο και μορφωμένο λαό που δεν έχει καμία σχέση με τον Λουκασέγκο και τους ε, ε, δικούς του. Σας ευχαριστώ κύριε ε, Τάνοκο. Ο κύριος Παλέτσκης είναι ο επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ε, απόφαση, χαιρετίζουμε την απόφαση να ελευθερωθούν οι 11 ε, πολιτικοί κρατούμενοι που είχαν κρατηθεί μετά τα γεγονότα της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Αυτή η απόφαση δεν είναι τυχαία σήμερα που συζητάμε ένα ψήφισμα και έχουμε την πρώτη συνεδρίαση της Euronest. Ε, είναι ένα πρώτο βήμα, δεν αρκεί όμως και θα πρέπει να καταδικάσουμε σαφώς την ε, ε, σύλληψη και τις καταγγελίες εναντίον του κυρίου Μπιαλέσκη και επίσης ο διάλογος θα είναι δυνατός μόνο μετά την ελευθέρωσή του και ε, αφού μας δοθούν στοιχεία για όλους τους πολιτικούς κρατομένους πρέπει να συντονίσουμε το μηχανισμό ε, στασίας προσωπικών στοιχείων σε ε, δικαστικές ε, διαδικασίες όταν έχουμε να κάνουμε με μη δημοκρατικά κράτη και παρακαλώ την Λευκορωσία να απαντήσει και να τεθεί και θέμα σχετικά με το κόστος των θεωρήσεων. Δεν είναι η πρώτη φορά που καταδικάζουμε το καθεστώ ε, στην Λευκορωσία που καταπιέζει του υποστηρικτέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανθρώπου από την κοινωνία των πολιτών. Καταδικάζουμε όμω τη στέρηση αυτή ελευθερία που αποτελεί ένα χαρακτηριστικό του καθεστώτος του Λασέγκο. Πρέπει να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο αυτή τη φορά. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται τα δικαστήρια όπως χρησιμοποιούνται τώρα. Εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε ο επικεφαλής ε, του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συνελήφθη στις 4 Αυγούστου 2011 να ελευθερωθεί και όχι να... Διακόπτει ο Πρόεδρος. Μιλάτε πιο αργά, παρακαλώ. Και είναι προφανές ότι το καθεστώς αυτό δείχνει πόσο μακριά μπορεί να πάει παραβιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συγχρόνως το καθεστώς δοκιμάζει τα όρια της δικιάς μας πολιτικής ευαισθησίας και ηθικής δέσμευσης. Εμείς Θέλουμε να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρη την κοινωνία της Λευκορωσίας. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να μένουν στην μοίρα τους στο καθεστώς ε, αυτό του Λουτασέγκο. Φτάνει πια. Το καθεστώς θα αναγκαστεί να συμμορφωθεί. Για να γίνει αυτό πρέπει να αντιδράσουμε στην αδικία αυτή που έχει γίνει ακόμα πιο ισχυρά από ό,τι το έχουμε κάνει κατά το παρελθόν. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι κατηγορίες κατά του Λιμπεράσκη βασίζονται σε ψεύτικα στοιχεία ε, που όπως λένε πήραν από την πολωνική τη λιθουανική κυβέρνηση βάσει διμερών συμφωνιών. Εγώ βέβαια δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της Πολωνίας, μπορώ όμως να μιλήσω ως Λιθουανός και ζητώ συγγνώμη για ό,τι έγινε στη Λιθουανία από τον Υπουργό Δικαιοσύνης εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως οι αρχέ τη Λευκορωσία εξακολουθούν να είναι υπεύθυνε. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσει το ψήφισμα αυτό και να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν από τέτοιε καταστάσει επειδή έγιναν κάποια τεχνικά λάθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει και θα ελευθερεί ο κύριο Μπλετσάσκη. Πρέντα είναι επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι χθεσινές εφημερίδες γράφουν σε πολλά μέρη της Ευρώπης ότι υπήρξε ε, μία πτώση του εθνικού νομίσματος της Λευκορωσίας κατά 40% κατόπιν της κρίσεως. Αλλά υπάρχει προγραμματισμένη οικονομία στη χώρα αυτή και αυτή η μέθοδος θα αποτύχει. Επίσης λέγεται ότι η ε, προγραμματισμένη ε, οικονομία ε, θα συνδυάζεται με καταστολή όπως και σε όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα και το, περίπου, το παράδειγμα του κυρίου Μπιαλέσκη είναι το τελευταίο που έχουμε. Πρέπει λοιπόν να αποφυλακιστεί και θα πρέπει να διαγραφεί από τον ποινικό κώδικα το άρθρο που λέει ότι δεν μπορεί κανείς ε, να συμμετέχει σε οργανώσεις. Ε, πρέπει ε, να, να αρνόμαστε τις θεωρήσεις στις χώρες αυτές και να παγώσουμε τα, τα περιουσιακά στοιχεία των ενδιαφερομένων. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ο κύριος Σόγκορ, μπορείτε να αρχίσετε από την αρχή και πάλι. Σας ευχαριστώ. Οι δραστηριότητες ε, ε, του κινήματος, ε, το οποίο ηγεί το ο Μπιαλάτσκι, το οποίο δημιουργήθηκε από το 1996, είναι υποδειγματικό για τη διάδοση της δημοκρατίας και την ανάδεση μιας κοινωνίας των πολιτών. Πρέπει να ενθαρρυνθεί να ενθαρρυνθούν και άλλοι άνθρωποι για να είναι τόσο θαραλέοι στις εκδηλώσεις τους και για να αναγκαστεί η Λευκορωσία να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θα πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε ότι κάθε εκφοβισμός είναι ίδιον της κάθε δικτατορίας ο πληθυσμός ε, θα βγάλει συμπέρασμα ότι είναι αδύνατο να νικήσει την ε, δικτατορία και να ξεφύγει από τα πλοκάμια της και γι' αυτό και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργήσει. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο πως η Λευκορωσία οφείλει να σεβέται τα... η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και αν δεν γίνει κάτι τέτοιο δεν θα μπορέσει να βασιστεί σε οποιαδήποτε υποχώρηση και συνεργασία από πλευρά των ε, χωρών της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα οι πολίτες πολίτες της θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη είναι στο πλευρό τους. Ευχαριστώ. Ρεπό, εκ μέρους των σοσιαλιστών παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ βλέπουμε ότι υπάρχει μία σκληρή καταπίεση ε, και διωγμός των δημοσιογράφων στη χώρα αυτή και μετά από τις προεδρικές εκλογές εκατομμύρια τόμων καταδικάστηκαν και ένας πολύ γνωστός ένα πολύ γνωστό άτομο είχε φυλακιστεί και αυτό είναι απλούστατα ένα παράδειγμα για το πώς ε, ε, προχωρά το κράτος αυτό ενώ ο καθένας θα έπρεπε να έχει δικαίωμα ελεύθερης ε, εκφράσεως. Ένα κράτος χωρίς διάλογο δεν είναι μία παραδεκτή κατάσταση. Πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος μέχρι ότου ελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι και γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο κύριος... Ε, τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μόλις επέστρεψα από την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης της Euronest που έλαβε χώρα, όπως γνωρίζετε όλοι, χωρίς τη συμμετοχή των λευκορώσων συναδέλφων. Κρίμα βέβαια για όλη την διαδικασία της Euronest, αλλά είναι ντροπή κυρίως για τον πληθυσμό της Λευκορωσίας. Και ένας είναι ο φταίχτης και αυτός είναι ο πρόεδρος Λουκασέγκο και το καθεστώ του. Πριν από μερικές εβδομάδες ε, ο ίδιος ο Λουκασέγκο υποσχέθηκε ότι θα ελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατούμενους. Αλλά αυτό που ήθελε είναι να προωθήσει την ε, οικονομία της χώρας, δηλαδή ό,τι κάνει πάντα. Και να που τελικά καταλήξαμε στη σύλληψη του Μπιαλάτσκι. Το κοινοβούλιο αυτό εξακολουθεί να πιέζει το καθεστώς του Προέδρου Λουκασέγκο ευτυχώς και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να το κάνει όσο δεν διαπιστώνουμε αλλαγές εκεί. Η απομόνωση όμως δεν φτάνει και το να καταδικάζουμε τον Λουκασέγκο. Όχι, πρέπει να βοηθήσουμε το λαό. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Μπίλαν από το ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η βίες ενέργειες και η σύλληψη του Αλές Μπιαλάτσκι προκαλούν την ε, οργή. Μας ε, εκπλήσει επίσης το γεγονός ότι οι πολωνικές και λιθωνικές αρχές εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς. Τα γεγονότα στην ε, Λευκορωσία δείχνουν ότι πρέπει πολλά να γίνουν. Χρειάζεται να λάβουμε σταθερή και έντονη θέση εδώ στις στις Βρυξέλλες απέναντι στη Λευκορωσία. Μπορούμε να συμβάλλουμε μόνο με αυτόν τον τρόπο στην αλλαγή της κατάστασης στη Λευκορωσία. Κάνω έκκληση στον κύριο Λουκασέγκο να απελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατούμενους. Καλό τις αρχές της Λευκορωσίας να νομιμοποιήσουν όλους τους κοινωνικούς οργανισμούς και να εγγυηθούν τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών της χώρας. Καλό επίσης όλα τα θεσμικά όργανα και όλα όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς να διευρύνουν και τις πιέσεις που ασκούν στις αρχές της Λευκορωσίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπίλαν. Η κυρία Βερζιά από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε οι στρατευμένοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίω η Γαλλική ε, Ένωση ε, την οποία εκπροσωπώ εδώ είναι πολύ ταραγμένη από την ε, σύλληψη του κυρίου και ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος αυτής της οργανώσεως. Ίσως ορισμένοι κοιτούν τα πράγματα στη χώρα αυτή με αποστερευρωμένη οπτική γωνία αλλά ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι άσχημη και επιδεινώνεται συνεχώς. Δεν μπορεί πλέον ε, να ε, λειτουργήσει μια μη κυβερνητική οργάνωση όπως η Βιάσνα και γι' αυτό ξεκίνησε ένα ε, λογαριασμό στο εξωτερικό και θεωρούνται αυτή τη στιγμή από τις αρχές της Λευκορωσίας σαν προσωπική η περιουσία του κυρίου Μπιαλάσκη και πρέπει ε, γι' αυτό να διωχθεί για φοροδιαφυγή ε, το οποίο δεν ευσταθεί αλλά ο κύριος Μπιαλάσκη έφτασε σε αυτή την κατάσταση λόγω της ε, μεταδόσεως πληροφοριών των αρχών από τις αρχές της Πολωνίας και της Λιθουανίας. Υποτίθεται ε, υπό το πρόσχημα της καταπολεμήσεως της τρομοκρατίας. Ε, καταδικάζω τις εμπλεκόμενες χώρες αλλά παρακαλώ κυρία Επίτροπε να πιέσετε τα κράτη να μην επαναληφθούν τέτοια περιστατικά και να μπορέσει να απελευθερωθεί ο κύριος ε, Μπιαλάσκη. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Πόσελτ. Κύριε Πρόεδρε, Ζητάμε να απελευθερωθεί ο κύριος Βιαλάσκη, ζητάμε μία ενισχυμένη στήριξη της δημοκρατικής αντιπολιτεύσεως και των ε, ελευθέρων συστημάτων στη Ρωσία και τέλος μία επιστροφή στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Δεν πρέπει ε, να ε, ξεχνάμε τι έγινε στην Νότιο Αφρική και ακόμη και σε ένα δικτατορικό καθεστώς μέσα στην Ευρώπη Γι' αυτό και στην τελευταία περίοδο ο κύριος Ντες με είχε στηρίξει να καταπολεμήσαμε και πολεμήσαμε κατά τρόπον ώστε να ξεχωρίσει κανείς τα δημοκρατικά δικαιώματα από τα θέματα της ανατολικής γυτνιάσεως και είχαν μπει όλα μαζί και δεν συμφωνώ γι' αυτό και είμαι ε, ευγνώμων στην πολωνική πολιτική η οποία ε, πέτυχε ε, στην διάσκεψη της ε, Πράγας το διαχωρισμό αυτό και τώρα που έχει την Προεδρία θα το βελτιώσει. Γι' αυτό χρειάζεται μία δημοκρατία στη Λευκορωσία κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αυτά τα συστατικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέρι. Ευχαριστώ. Η σύλληψη του κύριου Βιαλάτσκη στις 4 Αυγούστου στο Μίνσκ είναι άλλη μια απόδειξη τη κακή επίδοση στα ανθρώπινα δικαιώματα από πλευρά τη Λευκορωσία. Ο κύριο Βιαλάτσκι είναι κάποιο που αγωνίζεται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι αγωνιστή και η δουλειά του έχει συνεισφέρει υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για πολλού πολίτε στη χώρα του και με την κράτηση, η του έγινε ε, με το επιχείρημα ότι έχει διαπράξει οικονομικά αδικήματα. Αλλά αυτό είναι απαράδεκτο γιατί κατηγορείται ε, ότι κατηγορείται για κάποια αδικήματα τα οποία δέχεται το δικαστήριο χωρίς να είναι αλήθεια. Επιπλέον όμως αποτελεί και μια μεγάλη επίθεση σε βάρος της κοινωνίας των πολιτών. Πρέπει να θυμόμαστε, ο κύριος Βιαλάσκη είναι μία μόνο ακόμα περίπτωση ανθρώπου που διώκεται από τη Λευκορουσία ή άλλοι οι οποίοι είναι θύματα όχλησης από πλευράς του καθεστώτος. Θέλω και εγώ να ζητήσω την άμεση απελευθέρωσή του και αυτού και όλων των άλλων υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε για τον Μακή τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά και φαντάζομαι πως δυστυχώς δεν θα είναι και η τελευταία φορά που συζητάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Λευκορωσία. Η υπόθεση του κυρίου Άλες Μπιαλάσκη είναι ιδιαίτερη, ιδιαίτερα ανησυχητική και είναι ένα ακόμα παράδειγμα στη μακρά σειρά συλλήψεων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία. Ο κύριος Μπιαλάσκη, ο πρόεδρος του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι ε, μια απόδειξη για την ε, καταπίεση και την παρενόχληση των λευκορωσικών αρχών. Καλό ο Συμβούλιο και της Κομισιόν, καθώς και την είπα το εκπρόσωπο Κάθριν Άστον να μείνουν στις προσπάθειές τους για να καταδικάσουν τις παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία και για να υποστηρίξουν τους υποστηριχτές, το, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Επίσης καλώ τις αρχές της Λευκορωσίας να απελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και να σεβαστούν τις διεθνείς προδιαγραφές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γιατερμάκη. Ο κύριος Μαστάλκα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στηρίζω αυτούς οι οποίοι αποβλέπουν σε μια καλύτερη κατάσταση στη Λευκορωσία διότι όλοι πρέπει να σέβονται τις διεθνείς συνθήκες διότι έπρεπε να μπορεί κανείς να σέβεται τους νόμους. Δεν έχετε όμως το συνέστημα ότι αυτή είναι μία μονομερής προσέγγιση διότι πέρυσι υπήρξε ε, μία σύγκρουση μεταξύ ε, των Ισραηλιών με ένα ανθρωπιστικό άγημα και ε, φέτος υπήρχαν δύο οι οποίοι σκοτώθηκαν από κατά διαδηλώσει στην Αλβανία και τραυματίστηκαν άλλοι έξι ενώ ζητούσαν απλώς να προχωρήσουν σε εκλογές. Υπάρχει επίσης και ένας πόλεμος ο οποίος κηρύχθηκε εναντίον της Λιβύης. Ε, δεν έχετε το συνέστημα ότι εδώ υπάρχει μία οργανωμένη κίνηση κατά της Λευκορωσίας τη στιγμή που υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα και δύο τελευταία σημεία. Η, η, η ε, διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν υιοθετήθηκε το 1988 αλλά στο 10 ε, χρόνια αργότερα από ό,τι γράφεται σε, το, σε αυτό το ψήφισμα. Επίσης είναι πολύ ατυχές ότι δεν υπάρχουν πολλοί παρόντες σήμερα. Μία μπλε κάρτα από τον κύριο Πόσελτ. Κύριε, κύριε Μασάλκα, τη δέχεστε? Συμφωνείτε? Κύριε Πόσελτ, έχει το λόγο. Μία σύντομη ερώτηση στον κύριο Μαστάλκα. Δεν κατάλαβα την ομιλία του. Ήθελε δηλαδή να υπερασπιστεί τον δικτάτορα κύριο Λουκασέγκο. Θα ήμουν ε, ευτυχής εάν μπορούσαμε να μην υπερασπιζόμαστε μόνο αυτή τη διπλοπροσωπία και να έχουμε μία ενιαία αντιμετώπιση για όλα τα κράτη τα οποία αντιπροσωπεύουμε ε, και ε, για τα οποία συζητάμε. Μία μπλε κάρτα από τον κύριο Μπρέντα δεν είμαι βέβαιος εάν ο μιλητής δέχεται την ε, μπλε κάρτα μου. Τη δέχεστε κύριε Μαστάλκα. Μπορείτε να προχωρήσετε κύριε ε, Πρέντα. Αντιθέτως προς τον κύριο Πόσελ, το οποίος ε, ρώτησε το συνάδελφο αν υπεραμείνεται του Λουκασέγκο, εγώ θα ήθελα να ξέρω αν υπεραμείνεται και του Καντάφη. φοβάμαι ότι αυτοί οι οποίοι στο παρελθόν τον αγκαλιάζανε και ε, τον, ε, ε, τον υπερισφαζόντουσαν δεν φαίνεται τώρα να έχουν τώρα σχέση μαζί του. Ο κύριος Λίσκε, Λίσεκ. Κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο κύριος ε, Διαλάλσκι έχει συλληφθεί. Κάποιος ο οποίος πάντα αγωνιζόταν υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να υπερψηφίσουμε το ψήφισμα αυτό και να υιοθετήσουμε και άλλα στο μέλλον για την ίδια αυτή υπόθεση. Πρέπει όμω επίση να ξέρουμε ότι ο κύριο Λουκασέγκο κατά πάσα πιθανότητα δεν διαβάζει τα ψηφίσματά μα και ακόμα και αν τα διαβάζει δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία. Γι' αυτό πρέπει να υιοθετήσουμε μια άλλη αποφασιστική πολιτική από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να πούμε ξεκάθαρα στο Λουκασέγκο και στους συνεργάτες του, του αστυνόμους του, του δικαστέ του, όλους αυτούς να του πούμε ότι θα του θυμόμαστε, θα θυμόμαστε τα ονόματά τους. Δεν ξεχνάμε εκείνους οι οποίοι βάζουν στη φυλακή τους υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και έχω και μια παρατήρηση ακόμα όσον αφορά τις πολωνικές αρχές. Στην Πολωνία είναι ο Γενικός Αγγελέας ο οποίος τελικά ε, έδωσε τις πληροφορίες τις σχετικές με τον κύριο Βιαλάτσκι στις ε, αρχές της Λευκορωσίας. Η πράξη αυτή δεν έχει καμιά σχέση με τις πολωνικές αρχές. Το κοινοβούλιο μας, η κυβέρνησή μας έχουν καταδικάσει την πράξη αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε τώρα στη διαδικασία του Catch Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Κάλλη που έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η σύλληψη και η φυλάκιση στις 4 Αυγούστου του κύριου Άλες Βιαλάτσκη αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ίσως βέβαια να είναι το τελευταίο λάθος αυτού του δικτατορικού καθεστώτος. Γιατί οι άνθρωποι μετά και από την Αραβική Άνοιξη έχουν αρχίσει να ενθαρρύνονται και να αντιδρούν. Εφόσον λοιπόν έχει φυλακιστεί ένας τέτοιος υποστηρικτής ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξαιτία λένε οικονομικών αδικημάτων, εμείς πρέπει να αντιδράσουμε γιατί αυτό μπορεί να είναι μια δικαιολογία και μόνο. Δεν ισχύει. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε μια προθεσμία ώστε να βάλουμε και κυρώσεις στην χώρα αυτή εφόσον δεν προχωρήσουν απελευθέρωση του. Ευχαριστούμε ο κύριος Βόλσκι. Συμφωνώ με όλες τις ε, καταδίκες. Ε, είναι πρόβλημα ένας υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να τυχάνει τέτοιες μεταχείρισεις. Αλλά δεν είναι πρόβλημα ενός ανθρώπου. Σας παραθέτω την δήλωση της ε, συνέλευσης της Euronest που μόλις ολοκληρώθηκε σε μια άλλη αίθουσα εδώ και εγώ είμαι συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τη Λευκορωσία. Κάνει λόγο για τέλος των δίωξης των, αρχηγών της αντιπολίτευσης. Μιλά για τους κρατούμενος Μιλάει για 24, 24 ε, ακτιβιστές που οδήγησαν σε αναταραχές που κατέληξαν στην, στη φυλάκιση και άλλων ε, αντιρρησιών. Ε, καλούμε να σταματήσει η παρενόχληση, απειλές κατά της κοινωνίας. Ζητάμε να παγώσει η βοήθεια στο λευκορωσικό καθεστώς και ε, μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κρατούνται, οι δημοσιογράφοι και οι προεδρικοί υποψήφοι. Θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Το να σώσουμε έναν άνθρωπο δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά πιστεύω βέβαια ότι δεν θα σώσουμε ούτε αυτόν τον άνθρωπο γιατί ο Λουκασέγκο τι κάνει, αφήνει έναν και μετά πιάνει άλλους δέκα. Οπότε ε, τα πραγματικά αίτια βρίσκονται αλλού. Και θα ήθελα να σας πω επίσης ότι η συνέλευση της Euronest αυτό το ψήφισμα δεν το δέχτηκε, γιατί υπήρχε να ε, αντιρρήσεις εν γέννη από ευρωβουλευτές από πέντε χώρες και γιατί ήταν εξ εξαιρετικά δύναμη η παρουσία του σώματός μας. Δεν μπορούμε να μιλάμε εδώ, να ψηφίζουμε εδώ και να μην ενεργούμε και στα άλλα σώματα. Σας ευχαριστώ. Όμπερ Μάιερ. Κύριε Πρόεδρε, ο φυλακισμός του υπευθύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα κυρίου Μπιατλάσκη ε, και ε, έχει διευκολυνθεί με ε, την ατυχή βοήθεια που προσέφερε η Λιθουανία στο Λουκασέγκο ε, και η κίνηση του Μπιαλάσκη είχε υποβάλει, είχε καταθέσει χρήματα στη διπλανή χώρα και για τους λόγους αυτούς φυλακίστηκε. Μέχρι εδώ πάμε σχετικώς καλά, διότι ότι ίσως δεν έπρεπε να έχει καταθέσει το εξωτερικό. Αλλά ελπίζω ότι οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ ε, του Βίλνιους και της κοινωνίας των πολιτών δεν θα έχουν πληγεί από το γεγονός αυτό και ελπίζω ότι θα μπορέσει και ο, ο κύριος Μπιαλάσκη να έχει μία ε, αίσια έκβαση. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, δεν ξέρω πόσα άτομα ή πόσες ε, φορές εφέτος έχουμε συζητήσει την περίπτωση της Λευκορωσίας και τώρα ε, μιλάμε για τον κύριο Μπιαλάσκη ε, ο οποίος ήταν ο πρώην πρόεδρος του Κέντρου για Ανθρώπινα Δικαιώματα και ο οποίος κατηγορείται διότι απέκρυψε ε, χρήματα σε ένα τραπεζικό λογαριασμό στο Βίλνιους αλλά απλώ για να βοηθήσει τις δραστηριότητες της ε, οργανώσεώς τους δηλαδή ε, κατά των πολιτικών καταστολών. Επιπλέον αντιλαμβανόμαστε ότι η χώρα αυτή προσπαθεί να καταστήλει την ελευθερία στη χώρα αυτή και θα πρέπει να γίνει κάποια κίνηση κατά του καθεστώτος του Λουκασέγκο. Κύριε Πρόεδρε, ο, ο Αλέξανδρος Μπιαλάτσχη είναι ένας από τους γνωστότερους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορεσία. Είναι πραγματικά ε, εντυπωσιακό ότι διεθνείς διαδικασίε χρησιμοποιήθηκαν για να βοηθήσουν στη σύλληψή του. Βλέπουμε ε, ότι πρέπει να λαμβάνουμε προφυλάξεις με την ενημέρωση στις διαδικασίες ε, αίτησης δικαστικής βοήθειας σε διεθνείς ε, διαδικασίες. Ε, συνεργάζονται οι αστυνομίες, ε, συνεργάζονται οι δικαστικές αρχές, αλλά αυτή η συνεργασία δεν μπορεί να έχει κατάληξη, δεν μπορεί μάλλον να χρησιμοποιείται μέσα στο πλαίσιο παράνομων διαδικασιών που στόχο έχουν να συλλέξουν πληροφορίες για εκπροσώπους τη αντιπολίτευση, έτσι όπως έγινε για τον ε, Μπιαλάτσκι και ο συνάδελφος Λίσεκ είπε ότι ο Πολωνός εισαγγελέα που προέβη σε αυτή την πράξη ε, δέχτηκε κυρώσει στην Πολωνία. Πρέπει λοιπόν να, γίνεται σεβαστή, να γίνονται σεβαστές οι δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σαν τελευταίος ομιλητής σε αυτό το γύρο, ο κύριος ε, Γκάλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτά που μόλις είπε ο κύριος Σόνικ. Νομίζω ότι θα έπρεπε κανείς να περιμένει μία ε, πολιτική ευαισθησία από τις ε, εθνικές φορολογικέ αρχές όταν υπάρχει μία συμφωνία με μία δικτατορία. Και ελπίζω αυτό να το γνώριζαν όλοι. Και να είναι η τελευταία φορά που γίνεται μία τέτοια συζήτηση για κάτα ε, στολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στη Λευκορουσία και καλό θα ήταν να γίνει μια πιο ουσιαστική πολιτική γιατί μια πιο ουσιαστική συζήτηση για την πολιτική γυρνιάσεως με την ε, Λευκορωσία μια χώρα την οποία θα θέλαμε να καταλήξει σαν ε, δημοκρατικό καθεστώς. Είναι εδώ σωστό να τονίζουμε την κακή μοίρα ορισμένων συγκεκριμένων ατόμων διότι ορισμένοι θεωρούν ότι αναλαμβάνουν την κυδαιμονία ορισμένων περιπτώσεων για να ε, πλήξουν συγκεκριμένα καθεστώτα μέσω αυτών των ατόμων. Ευχαριστώ και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την περίπτωση του κυρίου Μπαλάση και η κυρία Μάλστραμ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί όλο ιδιαίτερω για την κατάσταση και για τι συνεχιζόμενε καταπιέσει σε βάρο τη κοινωνία των πολιτών, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωση και των υποστηρικτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευρά του Καθεστώτο. Η Κάθριν Άψον, η ύπατη εκπρόσωπο, έχει επαναλάβει πολλές φορές τις ανησυχίες της για τις εξελίξεις στη Λευκορωσία. Έχει καταδικάσει όλες τις πράξεις εκφοβισμού και όχλησης σε βάρος υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είπε ότι πρέπει να υπάρχει το καθεστώς ε, των μη κυβερνητικών οργανώσεων που υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Εμείς ζητάμε την απελευθέρωση του Άλες Βιαλάτσκι, υποστηριχτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ρόλο κλειδί στην κοινωνία των πολιτών στη Λευκορωσία. Κακός συνελήφθη με την κατηγορία της φοροδιαφυγής χωρίς να υπάρχει βάση σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει επίσης ότι πρέπει να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες έχουν, ε, οργανισμού, έχουν ε, λογαριασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες για να προστατευτούν ακριβώς από το καθεστώς πρέπει να συνεχίσουν να προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να καταγγέλλονται. Ο συνάδελφός μου, Επίτροπος Φιούλερ, τον Ιούλιο ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για να βοηθήσει τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις στη Λευκορωσία και σε επαφές με την αντιπολίτευση και με την κοινωνία των πολιτών εκεί. και αυτό στα πλαίσια μια συνάντηση συντονισμού με δωρητέ που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Συγχρόνως στηρίζουμε τον κύριο Μπιαλάτσκι όσον αφορά τα δικαστικά του έξοδα που είναι κάτι που αποτελεί μέρος ενός ε, ιδιαίτερου πακέτου που ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο στην Πολωνία ο Επιτροπός Φίλε. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να στηρίξουμε τον κύριο Βιαλάτσκι και άλλους πολιτικούς κρατούμενους και θύματα της καταπίεσης στη Λευκορωσία που είναι πολύ όπως είπατε και εσείς. Σημειώνουμε το γεγονός ότι απελευθερώθηκαν κάποιοι πολιτικοί ε, κρατούμενοι και την πρόθεση του Προέδρου ζήτηση Τρογγυλής Τραπέζης. Όμως ο διάλογος με την αντιπολίτευση στη Λευκορωσία πρέπει να ξεκινήσει εφόσον απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι. Εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τη Λευκορωσία ώστε να υπάρξει σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κράτου δικαίου και των δημοκρατικών αρχών στη χώρα. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να υψώνουμε τι φωνέ μα για να καταγγέλουμε του υπεύθυνου των ε, μέτρων ε, στέρησης ελευθερίας και θα στηρίζουμε την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να κινητοποιηθεί και η διεθνής κοινότητα ώστε να καταδικάζει και να καταγγέλει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, στη χώρα και στις 20 Σεπτεμβρίου στο Human Rights Council, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Επίτροπος θα μιλήσει για την κατάσταση αυτή στη Λευκορωσία και θα προτείνει ε, να δοθεί συνέχεια στο ψήφισμα που εγκρίνατε τον Ιούνιο εδώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μάλστρομ. Έτσι λίγη συζήτηση για την Λευκορωσία και θα ψηφίσουμε αμέσω μόλις έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για δύο ακόμα περιπτώσεις, η πρώτη από τις οποίες είναι το Σουδάν, η κατάσταση στο νότιο Κορδοφάν και τον Γαλάζιο Νείλο. Δίνω το λόγο ευθύ αμέσως για να ξεκινήσει η συζήτηση στον κύριο Τάνοκ.